Συνάδελφοι, σας παρακαλώ τις συζητήσεις σας εκτός της αιθούσης της Ολομέλειας και γιατί τώρα θα περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Κύριε Σάριος Βόλς και κύριε Τζιπ, κύριε Μπρόκ,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 Λοιπόν, φτάνουμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Η πρώτη ομάδα αφορά το σημείο 9 ή μάλλον 9 α, τέτοιου είδους α, επεξηγήσεις και θα σχετικά με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μορβάη. Στι χρηματοπιστωτικέ αγορές υπάρχουν ε, κάποια συγκεκριμένα πρότυπα και οι εκλογέ οι οποίοι με γνωρίζουν